Και υπάρχει διαδικαστικό από ένα συνάδελφο, ο οποίος θέλει να μας πει κάτι. Οπότε σας παρακαλώ, ησυχάστε για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. So please. Mr. Campbell. Παρακαλώ, κύριε Κάμπελ. Πρόεδρε, ναι, έχω διαδικαστικό. Όσον αφορά το άρθρο 130 για τις ερωτήσεις. Για το κόμμα μας είμαστε όλοι ευρωβουλευτές. Και το πιο σημαντικό δικαίωμά μας είναι να ελέγχουμε μέσω των, ερωτήσεων την εκτελεστική εξουσία. Οι ερωτήσεις όμως δεν παίρνουν τελικά κατάλληλες απαντήσεις, οι οποίες είναι υπεκφυγές συνήθως και πολύ συχνά δεν έχουμε καν απαντήσεις. Το άρθρο λοιπόν 130 σημείο 5 λέει έξι εβδομάδες είναι η προθεσμία για να απαντηθούν οι ερωτήσεις μας. Μερικές φορές όμως περιμένουμε 11 εβδομάδες για να έχουμε απάντηση. Οι τεχνοκράτες θα είναι γι' αυτό και είναι κάτι το οποίο υπονομεύει τη δημοκρατία, πρόεδρε. Πρέπει να αλλάξει τάχιστα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τα όρια αυτά εμείς τα έχουμε θέσει, μου υπενθύμησαν. Οπότε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το σημειώσαμε πάντως και θα μεταφέρουμε το σχόλιο σας στις αρμόδιες αρχές. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Λούνες. Μία ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Στη συνέχεια περνάμε στην έκθεση Τίας Τεμέρα Γκαρθία Κονσουέγρα. Τροπολογία αριθμός 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2. Διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Εγκρίθηκε λοιπόν έκθεση αυτή βάσει της Συμφωνίας ε, Κοινοβουλίου-Συμβουλίου. Σημείο 3 τώρα, έκθεση Βίλκστρομ. Εδώ έχουμε τις τροπολογίες 1 και 2 που είναι ίδιες, ταυτόσιμες. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. Η έκθεση εγκρίνεται βάσει της συμφωνίας ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και τώρα περνάμε στην πολιτική συνοχής. Έχουμε το σημείο 4 στο αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σημείο 6 αρχικού κειμένου. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία όμως. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Αιτιολογική σκέψη Β, αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία πάλι. Ψηφίστε παρακαλώ. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες και τώρα έχουμε τις επεξηγήσεις ψήφου. Συναδελφοί, έχουμε ακόμα επεξηγήσεις ψήφου. Να αρχίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, αρχίζουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Ντόλτεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Λόρδος Έμραϊ βοήθησε έτσι ώστε η Europol να γίνει ένα σημείο ανταλλαγής πληροφοριών πολύ πολύτιμο ανάμεσα στις νομικές αρχές. Σήμερα κάναμε ένα βήμα ακόμα στην καταπολέμηση